κάθε μέρα να συναντούμε. 10.000 πολίτες που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και που εκπροσωπούν εκατομμύρια ε, άλλων πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά, λέει ο Πρόεδρος. Κατατίθεται ψήφισμα πέντε ομάδων για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα έχουμε τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού δυνάμει το άρθρο 150 του κανονισμού με τον κύριο Τοκέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν από 91 χρόνια και ε, παραγνωρίζοντας ε, το δόγμα Wilson περί αυτοδιάθεση των λαών, η Τρανσιλβανία και άλλα μέρη της ε, Ουγγαρίας αποκόπηκαν από την πατρίδα μας χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των πληττόμενων των Ούγγρων, δηλαδή του πληθυσμού της περιοχής αυτής και πρέπει να πω ότι δεν θέλω να ανοίξω τώρα παλές ιστορίες ε, και ε, δαφικές διαμάχες, αλλά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να αφαιρεθεί από τον Ολιβέρ Μπορντόγια και μάλλον και από άλλους ε, συμπολίτε του η σλοβακική τους ηθαγένεια και να εκδιωχθούν από την πατρίδα τους στο Φέλβιντεκ της Σλοβακίας επειδή ε, προβάλλουν την ουκρική τους ταυτότητα. Είναι επίσης απαράδεκτο στην Τρασιλβανία της Ρουμανίας, στην πατρίδα μας, την πατρίδα μας, ε, στο δικό μας Ουγγρικό Πανεπιστήμιο του Μάρος Βαχάρσλη, Τύργου Μουρές τώρα, εμείς οι Ούγγροι να μην μπορούμε να ανοίγουμε τμήματα ουγγρικής γλώσσας και ιστορίας. Και επίσης όταν χάσαμε τα εδάφη μας, τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε και το δικαίωμα να προβάλλουμε διακόπητο, το μιλητής. Σμόλκοβα παρακαλώ. Na Στη Σλοβακία επικρατεί μεγάλη ε, αγανάκτηση γιατί απέτυχαν ε, τα όργανα τα οποία έπρεπε να τηρήσουν την ασφάλεια και η υπηρεσία πληροφόρησης και με την εισαγωγή ενός ε, ανίκανου πρώην υπουργού ένας δημοσιογράφος ο οποίος συμμετείχε και δούλευε στο Υπουργείο Άμυνας και το σκάνδαλο αυτό στα μέσα ενημέρωσης έγινε γνωστό και από υπηρεσίε που ασχολούνται με την ελευθερία του τύπου. Ελπίζω να γίνουν σχετικέ έρευνε προκειμένου σε ένα δημοκρατικό κράτο να μην επικρατούν τέτοιε ανασφάλειε για τα προσωπικά δεδομένα και για τι ε, δραστηριότητε και για την παρακολούθηση αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ο συνάδελφος Μπουσόη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Θεωρώ ότι έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα πρόοδου η Τουρκία. Την ενθαρρύνω να συνεχίσει τις προσπάθειές της και Παρά το γεγονό ότι παραμένουν αρκετά πράγματα που χρειάζεται να βελτιωθούν, θεωρώ ότι ο απολογισμό είναι θετικό. Ωστόσο, κάποια προσκόμματα που θέτει στο δρόμο τη Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω σε παραδείγματι το ζήτημα τη υποχρέωση για θεώρηση διαβατηρίων για του παρέχοντε υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και αποτρεπτικό βέβαια στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Υπάρχουν χώρε οι οποίε επιβάλλουν ποσοστώσει ω προ τα διακινούμενα από την Τουρκία φορτικά αυτοκίνητα, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο και με το πρωτόκολλο τη Άγκυρα, με την Συμφωνία τη Άγκυρα. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει, εφόσον η Τουρκία καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε από την πλευρά τη, να καταβάλουν και οι ευρωπαϊκέ χώρε. Αντίστοιχα, ευχαριστώ τον κύριο Μπούσο, η κυρία Ματίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απολογισμού όσον αφορά τις πολιτικές λιτότητες ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης, πολιτικές που έχουν επηρεάσει πολύ ε, πολλές χώρες, καθώς και για τις ε, διαρθωτικές υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις κοινωνικές συνθήκες όπου ζουν ένα σωρό κόσμος, όχι μόνο στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά και σε άλλα πλαίσια. Μόλις την περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία έγινε η μεγαλύτερη γενική απεργία που έχει γίνει ποτέ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά αν δούμε τους ανθρώπους που είχαν κατέβει στους δρόμους, βλέπουμε ότι είναι μια διαδικασία Βλέπουμε ότι κατέβηκαν στους δρόμους ε, και εδώ και στις Βρυξέλλες ε, την Παρασκευή προβλέπεται μεγάλη πορεία. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και τα αίτια των προβλημάτων είναι κοινά και γι' αυτό, χρειάζεται, και, γι αυτό και η αντίδραση του κόσμου είναι κοινή. Ευχαριστώ συνάδελφε Ματίας και τώρα ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι οι εκπρόσωποι της Σλοβακίας έχουν τρελαθεί με μια απόφαση της κυβέρνησης. Πολλοί γιατροί ε, καταναγκάζονται σε, εργασίες, σε εργασία, όπως στην εποχή του Χίτλερ και του Στάλιν. Η ελίτ των γιατρών εξαναγκάζεται με ποινή φυλάκιση και σε αντίθεση με τον εργασιακό κώδικα να δουλεύει μέρα νύχτα χωρίς να υπάρχουν ωράρια, όπως το επιθυμεί ακριβώς ο εργοδότης τους. Και η πολιτική αφήνει το θυμό τους να ξεσπάσει στους γιατρούς, στους γιατρούς εκείνους που θέλουν να αντισταθούν στην κυβέρνηση που θέλει να κλείσει τα τελευταία δημόσια νοσοκομεία. Κυρίε και κύριοι, πρόκειται για μια κατάχρηση τη δύναμη, τη εξουσία τη κυβέρνηση. Σήμερα είναι οι γιατροί. Αύριο θα μπορούσαν να είναι οι δάσκαλοι, οι, όλες οι εργασιακές τάξεις. Δεν είναι δημοκρατία αυτό πλέον, είναι δικτατορία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω και εκ νέου το θέμα της κινητικότητας των Ρουμάνων και Βουλγάρων ε, εργαζομένων, γιατί διοργανώθηκε μία συζήτηση για το θέμα αυτό υπό την παρουσία του Υπουργού Εργασίας της Ρουμανίας. Ε, καταδικάζουμε τις περιορισμούς που αποφάσισαν να παρατείνουν η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό καταστεί την κατάσταση πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη. Αδύνατη θα έλεγα για μας, γιατί θέτει υπερβολικά αυστηρά κριτήρια για την χορήγηση έγκρισης εργασίας οι Ρουμάνοι και οι Βουλγάροι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν καν αίτηση και αυτό αποτελεί διάκριση βάση εθνικότητας ενώ άλλες χώρες όπως η Ισλανδία άρουν τους περιορισμούς άλλες χώρες τις διατηρούν. Τι θα κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις 10 κρίσιμες ημέρες. Ευχαριστώ στον Αμπτουμπασέσκο και τώρα τα Μπάιντι. Στην Ευρώπη ισχύει από το ρωμαϊκό δίκαιο μέχρι σήμερα η απαγόρευση της ε, αναδρομικής ισχύω των νόμων. Όμως αυτό το παραβιάζει η Ουγγρική κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ε, πέρσι εισήγαγε νομοθεσία που τροποποιεί το ταξιδιωτικό σύστημα. 300.000 άνθρωποι πλήττονται από αυτές τις αλλαγές, οι οποίες είναι αναδρομικές. Από αυτό σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Και τώρα... Θέλει να επιβάλλει αναδρομική ισχύ και κάποιων τροποποιητικών διατάξεων ως προς το Σύνταγμα της Ουγγαρίας προκειμένου να καλέσει σε λογοδοσία την προηγούμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχοι ε, ενώπιον αυτή τη εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα κατά αυτή τη κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Ταμπάιντι. Γκάλαχαρ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Όταν κάνουμε μια προσπάθεια για να διασώσουμε το ευρώ, το κάνουμε διότι ξέρουμε πόσο σημαντικέ ε, θα είναι, πόσο δυσμενεί θα είναι οι επιπτώσει από την κατάρρευσή του για του πολίτε και για τι επιχειρήσει τη χώρα. Είναι πολλοί οι πολίτε που εργάζονται σκληρά σε όλη την Ευρώπη και στην πατρίδα μου βεβαίω, οι οποίοι ανησυχούν ιδιαίτερω για την αποταμίευσή του, για τα λίγα χρήματα που έχουν μπορέσει να συσσωρεύσουν αυτά τα χρόνια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εμπιστοσύνη και σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ αγορών και κοινού πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρε μέλη, θα πρέπει οι ηγέτε των χωρών μελών να αποκαταστήσουν αυτή την έννοια εμπιστοσύνη θεσπίζοντα ένα τείχο προστασία το οποίο θα ε, θωρακίσει το ευρώ. μια καλά συντονισμένη και ευπρόσδεκτη κίνηση από κοινού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Federal Reserve και την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πρέπει να ε, προχωρήσει και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την απόφαση. Διακόπτεται ο μιλητής. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ. Μάιερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκλογές στην ε, χώρα μου χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη απουσία του εκλογικού σώματος. Ε, μετράται στο 67-69%. Είναι μια συνταγματική διαδικασία η οποία δεν λειτουργεί και θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και την πολιτική γυτνίαση. Το κίνημα της 20 Φεβρουαρίου που ε, οδήγησε χιλιάδες ε, κόσμο στο Μαρόκο για να διαμαρτυρηθεί κατά του καθεστώτος ε, δείχνει ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει στάση θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τη στάση μας απέναντι στο Μαρόκο περί του οποίου ήταν ο λόγος μέχρι στιγμής Ευχαριστώ κύριε Μάιερ Νικολέσκου. Bună seara! Am dorit să intervin pentru a saluta rezoluția... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Βαλτική, στη συνάντηση των χωρών της Βαλτικής που έλαβε χώρα στην Εστονία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε το σχετικό ψήφισμα και ελπίζω να υποστηριχθεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας έχουν το χαμηλότερο επίπεδο πληρωμών. Τα, οι κράτη της Βαλτικής απαιτούν και υποστηρίζουμε αυτό το αίτημα να υπάρξει ένα δίκαιο σύστημα πληρωμών στην Γεωργία που θα αποτυπώνει τους όρους για τους γεωργούς σε όλη την Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατανομή των πόρων αυτών θα πρέπει να μην επιτρέπει διαφορές μεταξύ υψηλού και χαμηλού επίπεδου. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τα έτη 2014 και 2015. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Πλάμπ δεν είναι εδώ. Last Την περασμένη Παρασκευή ήταν η διεθνή ημέρα της κατάργησης της βίας κατά των γυναικών. Στην Ιρλανδία ε, ολοκληρώθηκε έτσι και η εκστρατεία 16 ημερών για το πέρας για την κατάργηση της βίας στα σπίτια. Καθημερινά στην Ευρώπη οι γυναίκες βιάζονται και δέχονται κακή μεταχείριση από τους συζύγους ή τους φίλους τους. Μία στις πέντε γυναίκες στην Ιρλανδία έχουν πέσει θύματα βίας στη ζωή τους, αλλά δεν υποφέρουν μόνο οι γυναίκες αλλά και τα παιδιά. Πέρυσι 1.600 ε, υποθέσεις εξετάστηκαν, από, μάλλον εισακούστηκαν από την ε, γραμμή βοήθειας ε, για την βία κατά των γυναικών στην Ιρλανδία. Εάν δε, λόγω της κρίσης κλείσουν τα ειδικά κέντρα, οι γυναίκες δεν θα έχουν πουθενά να στραφούν. Θα, θα πρέπει να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, αλλά δεν θα πρέπει να αφήσουμε τη λιτότητα να υποβαθμίσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σα ευχαριστούμε και τώρα η συνάδελφος Φιγκρέιδο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από την γενική απεργία τη 24η Νοεμβρίου, σήμερα το πρωί στην Πορτογαλία, χιλιάδε άνθρωποι τους οποίους κάλεσε η ΣΕΖΕΤΕΠΕ και άλλες συνδικαλιστικοί οργανώσεις και κοινωνικές οργανώσεις συγκεντρώθηκαν ε, στην πλατεία Δημοκρατίας στη Λισαβόνα ε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του προπολογισμού του κράτους του 2012 που υποτίθεται θα, θα από την πλειοψηφία με αποχή του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Διαμαρτύρονταν κατά των επιθέσεων στα δικαιώματα των εργαζομένων, μέσω των ε, μέσω της κατάργησης ε, διακοπών, την αύξηση της, ε, του ωραρίου εργασίας το εβδομαδιαίο κατά δύο ώρες, κατά διαφόρων επιθέσεων. Ε, επίσης αποφασίστηκε η συνέχιση του, του, του αγώνα κατά αυτή τη πολιτική που οδηγεί στην Πορτογαλία, την Πορτογαλία στο χάος. Επόμενη μεγάλη ε, μέρα θα είναι εβδομάδα ε, αγώνα. Στις 17 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει και ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φιγκεϊρίδου. Ο κύριος Διασμήρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι ότι ε, έχουμε μεγάλη εξάρτηση στον ενεργειακό τομέα από εισαγωγέ ε, κατά 90% του πετρελαίου, 60% του φυσικού αερίου. Έχουμε επίσης και στο, στον άνθρακα αντίστοιχη εξάρτηση. Άρα λοιπόν, εάν μειώσουμε την ικανότητα παραγωγής ενέργειας από, τα πυρηνικά μας, από τους πυρηνικούς μας αντιδραστήρες, θα ενισχύσουμε την εξάρτηση από τρίτε χώρε. η ενεργειακή στρατηγική έως το 2015 τίνει να εγκαταλείψει τη χρήση του άνθρακα. Το δε κλείσιμο των αντιδραστήρων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο σταδιακό και οργανωμένο, έτσι ώστε να μην ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εξάρτησή μας από τρίτα κράτη. Να μην επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διαστημίρο. Κυρία Τιτσέο. Σας ευχαριστώ, Ρουμανία. Αποτελεί ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο είναι ενωμένο. Είμαι ε, περήφανη που είμαι πολίτης της Ρουμανίας και όλοι οι πολίτες γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο χτες ε, διοργανώθηκε το συνέδριο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Συναμιλήσαμε για πολλά θέματα και σε ό,τι αφορά το μέσο για την ε, διασύνδεση της Ευρώπης δεδομένων των εξελίξεων στις υποδομές για τις μεταφορές θεωρώ ότι τα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν όσο πιο πολλές μετροπολικές ε, πολιτικές περιοχές γίνεται. Θα πρέπει να ενταχθούν επίσης στα δεκτία τέντη. το βιομηχανικό κέντρο Καλάτς θα πρέπει να καταστεί τέτοιο κέντρο, γιατί συνδέει το Δούναβι με την Κωνσταντσα και την Μαύρη Θάλασσα, τον πόντο Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ε, πολυεθνικό τέτοιο κόμβος και θα πρέπει να ενταχθεί και να δικτυωθεί με τις ειρηνικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ στην Αλφατικά και τώρα ο κύριος Μέρφη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ο Ντέβιτ Κάμερον μίλησε τη μαζική απεργία σήμερα ως ε, ανόητη ε, πράξη. Και αυτό από έναν εκατομμυριούχο που μιλάει για άλλους εκατομμυριούχους και προσπαθεί να υποσκελίσει, να υπονομεύσει δύο εκατομμύρια κόσμο που βγήκαν να απεργήσουν, να διαδηλώσουν κατά των πολιτικών λιτότητας της ε, κυβόρνησης. Το μήνυμα των απεργών ήταν σαφές σήμερα. Όσοι εδώ και μη παρέκει. Δεν θα πληρώσουν άλλο, δεν θα δουλεύουν παραπάνω για πιο χαμηλέ συντάξει, δεν θα ανοιχτούν άλλες περικοπές στους μισθούς και στι συντέξει και οι περικοπές ε, στο δημόσιο τομέα δεν θα γίνουν ανεκτέ. Θα πρέπει να σηκωθούμε λοιπόν και να ε, είναι σαφή η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας, που μπορούμε να έχουμε δύναμη στα χέρια μας. Ε. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβει δράση η εργατική τάξη και να βρεθεί αυτή η εξουσία. Ευχαριστώ συνάδελφε αδελφέ Μέρφη. Μισάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2004 Προσχώρησαν 10 νέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Αυτό έλπιζαν να ζήσουν. Άρα είναι απαράδεκτο σε μια ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διέκονται πολίτες μόνο και μόνο επειδή αποφάσισαν να ζητήσουν ένα δεύτερο διαβατήριο, όπως συμβαίνει στη Σλοβακία σήμερα το κοινοτικό δίκαιο περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που ξεπερνούν τις διεθνείς σχετικές διατάξεις. Παράλληλα αυτά, το κοινοτικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει τη διπλή υπηκότητα. Μάλλον, το κοινοτικό δίκαιο δεν ε, αναγνωρίζει τη διπλή αλλά δεν το αναγνωρίζεται η εθνική, στην εθνική νομοθεσία. Η διπλή υπηκότητα δεν μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα Ευχαριστώ, συνάδελφε Μίσαρο, Άλβες. Σας ευχαριστώ. Η κρίση μολύνει όλες τις, ε, όλα τα κρατημέλη και αυτά παίρνει διαστάσεις ε, άνευ προηγουμένου που επηρεάζει τις βασικές ε, ουσιαστικές δραστηριότητες των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων που ακόμα και αν είναι υγιείς οδηγούνται στην πτώχευση και στην εργαζόμενη τους στην ανεργία. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την οικονομία και την κοινωνία. Κανένας δεν δίνει σημασία στις βαθιές αναδιαρθρώσεις, στην περισσότερη λιτότητα περισσότερες αλλαγές που βραχυπρόθεσμα δεν, θα, δεν είναι ικανές να αναχαιτήσουν την πορεία της κρίσης στην Ένωση. Δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα, τα κρατικά χρέη και ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε στις επιχειρήσεις μας ε, ε, μια εξυγίαση. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερή και σίγουρη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ τον κύριο. Άλβες τώρα η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. το ζήτημα της ε, ηθαγένειας ρυθμίζεται με βάση την αρχή τη επικούρικότητα από τα κράτη-μέλη. Και ως απάντηση στην ε, τροποποίηση της νομοθεσίας ε, περί ηθαγένειας της Ουγγρικής Δημοκρατίας εισήγαγε και η Σλοβακία ένα νέο νομοθέτημα το οποίο επιδεινώνει πολύ την κατάσταση στον τομέα της ηθαγένειας. Ο Σλοβάκος πολίτης δηλαδή λαμβάνει από τις Σλοβακικές αρχές μια επιστολή βάσει της οποίας μπορεί να εκδώσει διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγηση και πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια εγκατάστασης ε, παραμονής δηλαδή στην ίδια του την πατρίδα. Πράγμα το οποίο αποτελεί σοβαρό ε, φραγμό στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Ε, ε τίθεται λοιπόν το ερώτημα σε ποιο βαθμό τέτοιου είδου παράλογα μέτρα είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης και του δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Σαββό παρακαλώ. Vă mulțumesc. Prin noua lege a sănătății, guvernul din România dorește Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ρουμανική κυβέρνηση θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα νοσοκομεία και να καταδικάσει έμεσα εκατοντάδες χιλιάδων Ρουμάνους πολίτες σε θάνατο. Τα νοσοκομεία πρέπει να βρίσκονται μέσα σε μια κοινωνία και να λειτουργούν για να σώζουν ανθρώπινες ζωές, όχι για να κερδίσουν χρήματα. Όμως, όταν είναι πολύ αραιή η κάλυψη σε εξειδικευμένους γιατρούς σε περιοχές της Επέθρου και ταυτόχρονα κλείνουν και τα νοσοκομεία που βρίσκονται εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί άνθρωποι αποστερούνται από την απλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται. Οι Ρουμάνοι είναι πάνω από 15 εκατομμύρια και δεν έχουν αρκετά λεφτά στη θέσή του, καθώ είναι φτωχό λαό, για να μπορούν να καλύψουν τοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πρόεδρε, ευχαριστώ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά μέσα που χορηγούνται σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, στη Ρουμανία. Μια αναπτυξιακή δηλαδή δυνατότητα την οποία τώρα γνωρίζουν οι Ρουμάνοι πολίτες που δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν μέχρι τώρα τα κονδύλια. Δεν είναι όμως γνωστά όλα τα, τα στάδια αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη, στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερες υπηρεσίες. μειώνοντας ε, τη γραφειοκρατία, διότι το κύριο πρόβλημα στην περίπτωση αυτή ε, και στη δυνατότητα για υποβολή ε, δικαιολογητικών για τέτοιου είδου χρηματοδότηση είναι πολύ, πολύ βαριά γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε την κατάσταση και να μειώσουμε την γραφειοκρατία προς τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας επισημάνω ένα περίεργο ε, φαινόμενο πολλοί συναδελφοί αναφέρθηκαν ήδη στην κατάσταση και την περιέγραψαν. Η κατάσταση λοιπόν είναι πραγματικά παράλογη και γι' αυτό είναι σημαντικό σήμερα το Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το επισημάνουν αυτό. Ένα Σλοβάκο υπηκό, ο Όλιβερ Πόλκοϊ, έχασε την υπηκότητα, δηλαδή την ηθαγένειά του, τη σλοβακική ηθαγένειά του, επειδή ε, έλαβε η ουγγρική υπηκότητα. Αυτό τι σημαίνει ότι στα μάτια της Σλοβακίας αποτελεί πολίτη άλλης χώρας και γι' αυτό λοιπόν θεωρείται περιττός. Τίθεται το θέμα του κατά πόσο μπορεί να επιβληθούν κυρώσει σε περίπτωση που ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί από τη γέννησή του, ε, ζει από τη γέννησή του στη Σλοβακία και πληρώνει φόρους, ε, έτσι απορριφθεί. Αποτελεί αυτό ε, παραβίαση του Σλοβακικού Συντάγματο, το οποίο ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί από τη Σλοβακική του δικότητα παρά τη θέλησή του. Το μέτρο λοιπόν αυτό πρόκειται για ένα τμήμα τη αντικριτική μεταχείριση των μειονοτήτων στη Σλοβακία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πέλτ, παρακαλώ. Οι οργανισμοί αξιολόγηση πιστοπιστικής ικανότητας είναι περίτη. Η Επιτροπή δεν ξέρει τι να κάνει, τελεί ένα μηχανία και ορισμένοι επίτροποι είναι ανεύθυνοι. Οι οργανισμοί επιστολιστικής αξιολόγησης ε, διατυπώνουν απόψεις, χαρακτηρίζουν, δίνουν βαθμολογία, επηρεάζουν ε, ή επηρεάζονται από το κλίμα που επικρατεί στις αγορές και όχι από μια γερή επιστημονική βάση για τις κρίσεις τους. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σε θέση να προξενήσουν δισεκατομμυρίων ευρώ ζημιά σε επιχειρήσεις ή χώρες. Δεν κάνουμε τίποτα όμως γι' αυτό εμείς εδώ. Πρέπει να αγωνιστούμε στην Ευρώπη για να διαφυλάξουμε την Ευρώπη, τα το ευρωπαϊκό συμφέρον. Υπάρχουν επίτροποι, υπάρχουν κράτη-μέλη που Υπάρχουν επίτροποι οι οποίοι θέτουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ελεύθερο τρόπο ορισμένα κράτη-μέλη και ουσιαστικά δρούν κατά τρόπο ε, εγκληματικό στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σόκορ, για να ολοκληρωθεί και η περίοδος αυτών των παρεμβάσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την αλλαγή της Σλοβακικής νομοθεσίας, ε, θεωρείται ότι χάνει ένα Σλοβάκος πολίτη την υπηκότητά του μετά την ανάληψη μια άλλη υπηκότητας. Πρόκειται για ένα περίεργο φαινόμενο Τώρα το θέμα είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ένας Σλοβάκος υπήκος, Όλιβερ Μπόλτοκι, από αυτόν τον πολίτη λοιπόν ε, στερήθηκε η σλοβακική του υπηκότητα παρά τη θέλησή του και θέλει λοιπόν ε, η σλοβακική κυβέρνηση να καταδιώξει όσους ε, επιδιώκουν να συνδεθούν με την η υπηκότητά τους με την προέλευσή τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίζουμε προκειμένου να μην οδηγούνται οι χώρες σε εντάσεις. Θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα αυτά και η Σλοβακία ακολουθεί σήμερα διαφορετικό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Σόγκορα, έτσι ολοκληρώνονται οι ομιλίε του ενό λεπτού. Ευχαριστώ του συναδέλφου που άκουσαν και του άλλου ε, συναδέλφους, να ευχαριστήσω τον, τον Επίτροπο που έμεινε μέχρι τόσο αργά. Ολοκληρώνεται λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση. Επόμενη, ε, ξαναξεκινάει η συνεδρίαση αύριο στις 8.30. Έχετε την ατζέντα και μπορείτε να την βρείτε και